πολιτιστικά αγαθά του Ιράν είναι στόχος ε, ε, στρατιωτικής επίθεσης. Ε, βέβαια έχουν ε, πολύ ταψιλή στρατιωτικό προπολογισμό οι Ηνωμένε Πολιτείε και κάπως θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να μην πάει χαμένο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο τώρα έχει ο Κύριε, Κύριε Πατεκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δούμε το Ιράν και το Ιράκ ως ε, κομμάτι μιας ευρύτερης εικόνας ε, για τη γενικότερη περιοχή. Βλέπουμε όλο και περισσότερα πολιταρχικά καθεστώτα να γίνονται πιο επιθετικά. Ε, βλέπουμε περισσότερη ανάμειξη στις υποθέσει ξένων κρατών, από σταθεροποίηση, βλέπουμε τι γίνεται, Ιράν, Ιράκ και σε άλλες χώρες όταν βλέπουν να μειώνεται η παρουσία παραδείγματος χάρη τον ΗΠΑ ε, αυτό μπορεί να δίνει ίσως ε, την αφορμή να είναι πιο επιθετικά κάποια καθεστώτα, αλλά υπάρχει και ένα κενό το οποίο πρέπει να καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης για να βοηθήσουμε να υπάρχει σταθερότητα και να αποφευχθεί το χάος ε, στην ευρύτερη περιοχή. Μιλήσατε στην ΑΦΕΤ ε, πάρα πολύ πιστικά, κύριε Μπορέλ. Είπατε ότι θα πρέπει να είμαστε ε, αυτοί οι οποίοι θα φέρουμε τη σταθερότητα ε, στην ευρύτερη γειτονία. Αν θέλουμε να είμαστε πιστικοί και νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε πράξη αυτό τώρα. Σάντος, για ένα λεπτό, είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Στι αρχέ του έτου, η Μέση Ανατολή χαρακτηρίστηκε από την ανεύθυνη και μονομερή συμπεριφορά των ΗΠΑ και με την εξοδικαστική εκτέλεση του στρατηγού Σουλημανή. Κολοσιαίο λάθος, μνημειώδες σφάλμα των ε, Ηνωμένων Πολιτειών που θέτησε κίνδυνο και την πυρηνική συμφωνία από την οποία απαχώρησαν οι Αμερικανοί. Βέβαια αυτό δεν είναι το πιο επίγον. Ε, ε, η ε, κατά λάθο ε, κατάρρευση του ουκρανικού αεροσκάφους από την Τεχεράνη ε, οδήγησε σε μια κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να προωθήσει το διάλογο, να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει και να κατεβράσει τι εντάσει και να προσπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει το Ιρανικό καθεστώ να σταματήσει να καταπιέζει του ειρηνικού διαδηλωτέ που ζητούν μεταρρυθμίσει. Η γεωπολιτική κατάσταση δεν επιδέχεται διστακτικότητα και ενδιασμούς. Και γι' αυτό χαιρετίζω την απόφαση της Παρασκευής να ενισχυθεί η εντολή του υποτεκπροσώπου και να προσπαθήσουμε να σώσουμε την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, γιατί δυστυχώς ε, καθυστέρησε πολύ η εφαρμογή της και είναι σημαντικό για την περιοχή και για τον κόσμο να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και ενότητα και την απαραίτητη αποφασιστικότητα για να προσπίσουμε αυτή την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Ευχαριστώ. Ας ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, τα πρόσφατα γεγονότα σε Ιράν και Ιράκ μας δείχνουν πόσο εύθραυστη είναι σταθερότητα στον κόσμο. Και ποτέ δεν είναι μακριά η κλιμάκωση. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στον κόσμο. Πρέπει να μιλούμε όλο και περισσότερο με μία με ενιαία φωνή. Θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτέ δυνατότητε. Είναι καλό που θέλουμε να παραμείνει ζωντανό το πυρηνικό πρόγραμμα. Πρέπει όμω να προειδοποιήσουμε το Ιράν. Οι Ιρανοί διαδηλωτέ δεν πρέπει να ε, είναι άνθρωποι οποίοι θα πάθουν το παραμικρό. Καλό τον ύπατο εκπρόσωπο να διπλασιάσει προσπαθίες του και να αρχίσει ε, αυτός ο διάλογος μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν που είναι η μόνη λύση για να βγούμε από το διέξοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα κύριος ε, Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πατεκπρόσωπε, να ξεκινήσω με ένα ρεαλιστικό σχόλιο είναι αδύναμο ε, το ευρωπαϊκό χέρι. Έχουμε ένα μικρό ρόλο. Αν όμως θέλουμε να λάβουμε σοβαρά τις ευθύνες μας, ε, ε, θα πρέπει να συντονιστούμε. Αυτός ο συντονισμός θα πρέπει να είναι στα χέρια τα δικά σας, γιατί αυτή είναι και η αρμοδιότητά σας. Κύριε Μπορέλ, θέλουμε το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση να το υποστηρίξουμε. Ταυτόχρονα όμω ξεκάθαρα ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, την, ε, Ιρακινή, την Ιρανική καταπίεση και καταστολή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, την έκκληση για το Instex. Θα πρέπει να ε, γίνουμε εταίροι, πρέπει να προσχωρήσουμε και να βάλουμε και χρήματα στο Instex. Και το τελευταίο που θέλω να πω εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλά ε, σύννεφα, μαύρα σύννεφα, αλλά υπάρχει και κάτι θετικό που είναι οι Ιρανοί και οι Ιρακινοί πρόσφατα πολίτες που διαδηλώνουν. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό, κυρία Κέμπα. I'm sorry. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, ε, λάθος μου, προηγείται το κύριος Μάγερ, μετά η κυρία Κέμπα. Κύριε Μάγερ, έχετε ένα λεπτό συγγνώμη. Ευχαριστώ κύρια πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτό που βιώνουμε νομίζω εδώ είναι ε, ένα παιχνίδι ε, πολύ εγωιστικό και πολύ επικίνδυνο. Και οι δύο πλευρές ε, εγωπαθώς κυνηγούν τους στόχους τους. Στις ίπα ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία για την τρομοκρατία. Και στο Ιράν λένε πρέπει να παραμείνουν ήσυχοι οι διαδηλωτές. Και τελικά τι γίνεται στη μέση, τι υπάρχει. Ένα ουκρανικό αεροσκάφος το οποίο καταρρύπτεται. Τι βλέπουμε να γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες είχε αυτόν τον Νοέμβριο ε, να ζήσει ο ε, Τραμπ και τους αρέσει των Αμερικανών όταν κάποιος ε, με στιβαρό χέρι υποτίθεται αντιμετωπίζει την τρομοκρατία. Επίσης, το Ιρανικό καθεστώς χρειάζεται την αλληλεγγύη των πολιτών του, αλλιώς δεν πρόκειται να παραμείνει έτσι σε, στην εξουσία αυτό το αντιδημοκρατικό καθεστώς. Ευχαριστώ. Κύριε Μάγερ, δέχεστε το κύριο Μπουτικόφερ μπλε κάρτα. Κύριε Μπουτικόφερ, κύριε Μάγερ, σε σχέση με την κατάρριψη ε, του Ουκρανικού ε, αεροσκάφους. Ε, ουσιαστικά μιλήσατε για ατυχία. Υπήρξαν άμαχοι. Νομίζω πρέπει να στήσετε συγγνώμη γι' αυτό. Δεν μπορεί κανείς να και στη μέση αυτό το κρανικό αεροσκάφος και κατερρύφθηκε. Δηλαδή ήταν κάτι τυχαίο και κρίμα. Γιατί είναι πολύ κοινικό αυτό. Να έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Μάγερ, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβετε καταλάβετε ότι εγώ αυτό που έλεγα, έλεγα ότι είναι τυχαίο και καταλαβαίνετε πώς το εννοούσα και μην χρησιμοποιείτε τα λόγια μου, μην χειραγωγείτε αυτά τα οποία είπα. Και έπαγε ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Αλλά δεν χρειάζεται να κραυγάζουμε για υπεροψία και αλαζονία. Ε, μέχρι στιγμή, βέβαια, δεν μα γεμίζει αισιοδοξία η συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλού μηχανισμού και πολλέ δυνατότητε και ευκαιρίε, όχι μόνο διπλωματικέ, αλλά και αναπτυξιακή ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση δείχνει ιδιαίτερα στο Ιράκ ότι οι στρατιωτικές αποστολές, ιδιαίτερα του ΝΑΤΟ και των συμμάχων που θέλουν να αποχωρήσουν από την περιοχή αυτό, αυτή η, πρόθεση αποχώρησης είναι ανεύθυνη γιατί χρειάζεται σταθεροποίηση το Ιράκ και οι εντάσεις με το Ιράν δημιουργούν μια πολύ δύσκολη και έκριθμη κατάσταση. Είχαμε ψήφισμα για την κατάσταση των Γεζιντή. Η κατάσταση και των χριστιανών, χριστιανικών μειονοτήτων είναι δύσκολη. Ε, τι θα γίνει, θα γυρίσουν οι Γεζιντή. Ε, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε να υπερψηφίζουμε ε, τέτοιο περιεχόμενο ψηφισμάτων. Αυτό είναι ανάρμοστη συμπεριφορά. Και φαίνεται ότι στη Ρική Ανατολή η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ απόμακρη δυστυχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριος Μποτενγκά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ο Ντόναλτ Τραμπ εκφοβίζει αυτή τη στιγμή και πρώτους από όλους και τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι ε, για τέσσερις ημέρες ε, στο Twitter, στο διαδίκτυο, βλέπαμε το hashtag «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Το συνειδητοποιείτε αυτό και εσείς δεν μπορείτε καν να καταδικάσετε τη δράση του. Λέμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα. Ξέρετε όμως ότι ενεπλάκησαν ήδη στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία και στο Λίβανο οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε τι καταστροφή προκάλεσαν εκεί πέρα. Θέλετε και άλλη καταστροφή και άλλη παρέμβαση καταστροφική των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά δεν ρωτάτε κανεί σε ποιο πλανήτη ζείτε. Αν θέλετε λοιπόν να διασφαλίσετε, να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, ασχοληθείτε λίγο με τη στάση του ΝΑΤΟ. Αν θέλετε λοιπόν να προασπίσετε τους Ιρακινούς πολίτες θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Ιρακινού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να σταματήσουν προφανώς οι κυρώσεις οι οποίες στρέφονται κατά του ίδιου του Ιρακινού πληθυσμού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Πάτεν έχει το λόγο. Πριν από τα Χριστούγεννα είχα πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα με το Ιράν, το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, έπνε τα λίστια και ότι χρειαζόμασταν ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο. Κύριε Μπορέλ, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι τα όσα είχα πει τότε αληθεύουν, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται και συντοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση δεν προωθεί την ειρήνη, το αντίθετο κάνει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εγκαταλείψει το σχέδιο αυτό. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να προωθούν την δραστηριότητα των φυγκοκεντριτών ουρανίου οι δυνάμει του Ιράν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή τη στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να επέμβουμε επικοδομητικά στο Ιράν. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να παρέμβουμε μέσω της Ουάσιγκτον. Το εναλλακτικό λοιπόν αυτό σχέδιο θα πρέπει να έχει και την ίδια τη σύμφωνη γνώμη του Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις διαντιπροσώπων κατά των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και θα πρέπει έπειτα μέσω του εμπορίου να αναστήσουμε τις σχέσεις που έχουμε με το Ιράν. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο μέσω των οικονομικών σχέσεων μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα επιτυχές συναλλακτικό σχέδιο έναντι του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράση και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την ειρήνη στην όλη περιοχή. Ο κύριος τον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωπε. Την ε, περασμένη Τετάρτη το ουκρανικό αεροσκάφος καταρρίφθη και 176 ε, επιβαίνοντες ε, έχασαν τη ζωή τους. Η σκέψη μας πηγαίνει προς τα θύματα και τις οικογένειές τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. 18 μάλιστα από τους επιβάτες ήταν Σουηδοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταδικάσει απερίφραστα αυτή την ενέργεια του Ιράν και να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για την διαλεύκαση της υπόθεσης. Επίσης, οι υπέτοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Οι οικοί των θυμάτων έχουν δικαίωμα στην αλήθεια και επίσης δικαιούνται και αποζημίωση οι οικογένειες των θυμάτων. Επίσης, οι ε, Διαδηλώσει και διαμαρτυρίες κατά του Ιρανικού καθεστώ αποκτούν όλο και μεγαλύτερε διαστάσει. Θα πρέπει λοιπόν αποφασιστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τι δημοκρατικέ δυνάμει στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε κυρία Γκούτελαντ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, η ασφάλεια στο Ιράν και στο Ιράκ ε, κινδυνεύουν, κινδυνεύει. Ε, βρισκόμαστε στο χείλος ενός πιθανού πολέμου και η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Πολιτειών και Ιράν ε, έχει πάρει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στο Ιράν ότι θέλουμε ένα ειρηνικό δημοκρατικό μέλος με σεβασμό, μέλλον με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τήρηση της συμφωνίας για τα πυρηνικά. Την περασμένη εβδομάδα καταρρίφθηκε ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας της Ουκρανίας με 176 επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους. Και αιτία αυτής της τραγωδίας ήταν η κλιμάκωση της έντασης. 17 μάλιστα θύματα είτε ήταν Σουηδοί υπήκο, είτε, είτε είχαν σχέση με τη Σουηδία. Ήταν νέοι και παιδιά τα θύματα αυτά. Θα πρέπει να απαιτήσουμε λοιπόν τη διεξαγωγή εξονυχιστική έρευνα και θα πρέπει οι ενδιαφερόμενε χώρε να εμπλακούν στην έρευνα αυτή. Τα οικογένει, οι οικογένειε των θυμάτων δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια και επίση δικαιούνται αποζημιώσει. Θα πρέπει να γνωρίσουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί συνέβη αυτό το τραγικό γεγονό. Σα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Πόριτ. Κύριε Πίτροπε Μπορέλ, βλέπουμε ότι μέσω όλων αυτών των εντάσεων που έχουμε μεταξύ Ιράν, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι διαμεσολαβητή. Οποιασδήποτε επαφέ έχετε αυτή τη στιγμή με το Ιράκ θα πρέπει να, έχουν να κάνουν με την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε οι οποίοι αυτή τη στιγμή α, κρατώνται α, παράνομα από το Ιράν, όπω η κυρία Ράτκλιφ που έχει περάσει τέσσερα χρόνια στην φυλακή στο Ιράν και είναι από τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Καταλαβαίνετε φαίνεται ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εχθρική αυτή στάση του Ιράν απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συναντηθείτε και με μένα και με τον κύριο Ράτσι, το οποίο βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό, αλλά και οι, υπόλοιπες, ε, οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των οικογενειών, των ανθρώπων εκείνων που βρίσκονται παράνομα σε φυλακές στο Ιράν θέλουν να σας συναντήσουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να διαπραγματευτούμε την κατάστασή τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει προφανώς να απελευθερωθούν, διαφορετικά δεν μπορούμε να εγκρίνουμε και να προωθήσουμε καμία άλλη συμφωνία με το Ιράν στο μέλλον. Για ένα λεπτό, κυρία Γκρεγόροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ειρηνικούς διαδηλωτές στο Ιράν. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δέχονται διάφορες δράσεις καταστολής και αυτές θα πρέπει προφανώς να καταδικαστούν από μας. Η ε, στρατηγική αυτή τη στιγμή των ε, Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα στη Λιβύη, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, στο Ιράν. Έχουμε πολλές αποτυχημένες παρεμβάσεις από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρετε ότι η χειρότερη επιλογή μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τα καθεστώτα μέσω στρατιωτικής παρέμβαση. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στου Αμερικανού. Μην αποσταθροποιείτε περισσότερο την περιοχή αυτή. Θα πρέπει προφανώ να προωθήσουμε πολύ περισσότερο περισσότερο διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές συμφωνίες. Κύριε Μπορέλ, ξεκαθαρίστε το αυτό προς το Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υποστηρίξει καμία στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Ανταυτού θέλουμε μία συνεργασία οικονομική που θα προωθήσει όσο δυνατόν περισσότερο στι εμπορικέ μα σχέσει, αλλά και τι ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων στο Ιράκ. Η κυρία Σαρντών έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό όσον αφορά την κρίση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και όσον αφορά την επέμβαση στο Ιράκ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι κατακαιρματισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι ταχθήκαμε με το Ιράν μόνο και μόνο για να αντιταχθούμε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Για πάρα πολλές μέρες όμως είδαμε ότι σε ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ο στρατηγός Σουλεϊμανή θεωρήθηκε ήρωας. Ας μην ξεχνάμε όμως τι έχει κάνει το ίδιο το Ιράν. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι το Ιράν αυτό το οποίο κατέριψε το αεροσκάφος των Ουκρανικών αερογραμμών με 176 θύματα. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαμαρτυρίε αυτή τη στιγμή κατά του καθεστώτος του Ιράν. 1.500 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια στο Ιράν. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταλήξει στι φυλακές, έχουν αποτελέσει θύματα βασανιστήριων. Το ίδιο ισχύει και για πάρα πολλέ γυναίκες στη χώρα αυτή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή Χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μια Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αυτή τη Φεντερίκα Μογκερίνη, η οποία είχε το θράσο να πάει πριν από μερικά χρόνια στο Ιράν, προωθώντα συμφωνίε και χωρί να καταδικάζει καθόλου την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώ αυτή τη χώρα. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Now for one minute, Mr. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριο Κούλογλου. Κύριε Μπορέλ, με εξέπληξε λίγο η ομιλία σας γιατί ξεχάσατε κάποια πράγματα. Ποιο δολοφόνησε ποιον. Ο κύριος Τραμπ δολοφόνησε τον κύριο Σουλεϊμανί. Ποιο το ενίσχυσε με τις δολοφονίες ε, και τις ε, κυρώσει, ποιο ενίσχυσε τους σκληρού τη Τεχεράνη. Ο κύριος Τραμπ. Έχω το προνόμιο να κατάγομαι από μια χώρα με τον μόνο πρωθυπουργό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στήριξε ανοιχτά την δολοφονία πέρα από τον κύριο Τζόνσον και βεβαίως τον κύριο Νετανιάχου. Οπότε αυτό το οποίο θέλω να σα πω είναι ότι βεβαίως πρέπει να πιέσουμε το Ιράν να σεβαστεί τη συμφωνία και να παραχωρήσει δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά να ασκήσουμε και πίεση στο ΣΥΠΑ. Αλλιώ ο κύριος Τραμπ μας θεωρεί δεδομένο κύριε Μπορέλη. Σα Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντλ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τέσσερις σύντομες σκέψεις. Το πρώτο είναι τι διακρίνει τις ΗΠΑ από το Ιράν. Τι είναι το Ιράν, τι σημασία έχει αυτή η πυρηνική συμφωνία για μας σήμερα και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΗΠΑ είναι μια αρχαία δημοκρατία η οποία λειτουργεί. Το Ιράν είναι ένα πολιταρχικό καθεστώ το οποίο παραβιάζει συνεχώ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μου προξενεί έκπληξη το ότι και σε αυτήν την αίθουσα από του αριστερού και ε, δεξιού λαϊκιστέ αξισώνονται οι δύο χώρε. Είναι όμω και ένα υποκείμενο του διεθνού δικαίου το Ιράν, με το οποίο έχουμε μια διεθνή συμφωνία, την πυρηνική συμφωνία. Είναι σημαντικό αυτό για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και ακριβώς τώρα απειλείται αυτό ο μηχανισμός επίλυση διαφορών. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το οποίο πρότεινε ο Αυστριακός υπουργό Εξωτερικών, δηλαδή μια διπλωματία ενδιάμεσου μεταξύ Ιράν και ΙΠΑ, γιατί οπωσδήποτε οι συνομιλίες είναι καλύτερες από τους πυροβολισμού. Και βεβαίω νομίζω ότι καλύτερο θα είναι ε, εμείς να παίξουμε αυτόν τον ρόλο του ενδιάμεσου κύριε Μπορέλ. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Κώστα. Βασικός υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση στην ε, Μέση Ανατολή είναι η δικτατορία των Αγιατολάδων. Ο Σουλεϊμανί είχε σχεδιάσει και εκτέλεσε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Ήταν υπεύθυνο για την βία ή καταστολή των διαμαρτυρίων γενναίων Ιρανών πέρσι για ελευθερία και δημοκρατία οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους. Το Ιρανικό καθεστώς είναι ομοφοβικό και αντισημιτικό. Έχει ως ρητό στόχο την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποφασισμένοι εναντίον του. Η δολοφονία Σουλεϊμανή είναι αμφίβολη σύμφωνα με το διεθνές πολιτικό δίκαιο. Δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη με περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή της διπλωματίας. Πρέπει να σώσουμε την πυρηνική συμφωνία. Πρέπει η κυβέρνηση Τραμπ να έρθει να επιλύσει τις διαφορές σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Εμείς λοιπόν είμαστε στο πλευρό των διαδηλωτών που θέλουν ένα κοσμικό Ιράν και παλεύουν για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. De, de nous demander que faire, voyons la nouvelle réalité proche-orientale. Le régime iranien est désormais aussi contesté sur son sol qu'au Liban et qu'en Irak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 Βλέπουμε ότι η Ρωσία και πάλι βρίσκεται μόνη τη ε, στην ε, Μέση Ανατολή την ίδια στιγμή που ε, χάνονται οι δυνάμεις της στη Λιβύη. Διαχέονται οι δυνάμεις της Μανού. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Ιράν ή από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ah <laughs> c'est maintenant, donc euh, désolé si vous pouvez répéter. Excusez-moi. Εντάξει, λειτουργεί η διερμηνία. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ξεκινώ από την αρχή. Πριν αναρωτηθούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, α εξετάσουμε την πραγματικότητα στην Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό καθεστώ αμφισβητείται και στην επικράτεια, καθώ και στο Λίβανο και στο Ιράκ. Και η τραγωδία του Ουκρανικού Boeing έχει αυξήσει ε, την κριτική εναντίον του, ακόμα και στο εσωτερικό τη επικράτεια. Η αμφισβήτηση ε, της θεοκρατίας ε, αποδυναμώνει και τον ISIS ενώ βλέπουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις διαχέονται ε, αλλού. Τι μπορούμε λοιπόν, να κάνουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τις ΗΠΑ ή το Ιράν να αλλάξει η πορεία. Δεν μπορεί να επιλύσει αυτή την κρίση, αλλά μπορούμε να ε, απο, αποστείλουμε το μήμα προ όλου ε, όσοι έχουν υπογράψει την πυρηνική συμφωνία και προς τον Ασάτ και προς τη Ρωσία ότι πρέπει να βρεθεί μια περιφερειακή ε, συμβαστική λύση, αλλιώς θα βρεθεί ε, μόνη της. Merci. Now for one minute. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Χάν. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, η στοχευμένη δολοφονία ανθρώπων είναι βαρβαρότητα, όπως επίσης και η απειλή να καταστραφούν πολιτιστικά μνημεία η δολοφονία του Σουλεϊμανί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε γίνει από ειδικοί στον πόλεμο, ειδικοί στην ειρήνη και χάρη στη ΣΥΠΑ. Και γνωρίζουμε πως η πολιτική αποτυγχάνει όταν δεν τηρεί κάποιες αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να τηρείται το διεθνές δίκαιο ή συμφωνίες στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και αυτό περιλαμβάνει και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Αυτό το οποίο μετράει δεν είναι America First και Europe First, αλλά ότι μαζί ε, είμαστε όλοι. Δεν έχουμε χρόνο να ξεχάσουμε τα διδαχτήματα του παρελθόντος. Χρειάζεται ειρήνη αντί για πόλεμο. Χρειάζεται μια κοινή διατλαντική πολιτική που θα βασίζεται σε κοινέ αξίες ή τουλάχιστον κοινού στόχους σε γεωστρατηγικά ζητήματα για το περιβάλλον και το κλίμα, γιατί το ρολόι είναι στο παραπέντε. Μόνο ενωμένοι είμαστε μαζί. Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη και για την διατλαντική σχέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Τόματς. Ναι, κύριε Τόματς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι η δολοφονία του Σουλεϊμανή αποτελεί βάρβαρη πράξη. Θεωρείτε ότι είναι ε, πολύ λίγο το να εξολοθρευτεί ένας τρομοκράτης. Είναι τρομοκράτης ο κατά την, ε, κατά την αποψή σας ή όχι. Now, Mrs. Κυρία Χάν, για 30 δευτερόλεπτα έχετε το λόγο. Ich Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι ε, είχαμε μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τώρα, εμείς δεν θα κάνουμε το δικαστήριο εδώ μέσα. Λοιπόν, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και είναι σαφές. Αυτό και πρέπει να το πούμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χακαράινεν, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το Ιράν ε, που κυβερνάται από τους Ισλαμιστές είναι η κύρια απειλή στην ε, περιοχή. Το Ιράν ε, έχει διασκορπίσει παντού το στρατό του στην περιοχή. Το Ιράν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο αυτό σε καμία περίπτωση και ο δεύτερος στόχος θα είναι να καταστρέψει το Ισραήλ. Συνεπώς, ε, η προσφυγή στα πυρηνικά όπλα, η κούρσα μάλλον, ε, είναι κάτι που βλέπουμε στην ε, περιοχή και δεν θα κάτσει το Ισραήλ με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει η Ευρώπη να σταματήσει να ανακατεύεται, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι εφικτό. Όταν θα εξαντληθούν τα πετρέλαια, δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζόφκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους ε, είδαμε ε, απρόσμενα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και αλλού με 3.000 στρατιώτες από 19 κράτη-μέλη. Τα γεγονότα αφορούν και την ασφαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση στο Ιράν και στο Ιράκ είναι ιδιαίτερα ενισχυτική και, είναι, και καλωσορίζουμε τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Καλό μέρη που εμπλέκονται να δώσουν χώρο στο διάλογο. Πρέπει να βοηθήσουμε του εταιρείε μα για να ανοίξουν διπλωματικού διάβλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπίσει το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση και να πείσει το Ιράν ότι είναι προ όφελό του να σεβαστεί αυτή τη συμφωνία. Επίση, η σχέση με το Ιράκ πρέπει να είναι παραγωγική και σταθερή. Αφού ε, υπέφερε ε, η χώρα από το ISIS, τώρα βρίσκεται υπό ανοικοδόμηση. Πέρσι ήμουν εκεί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ στη Βαγδάτη και πραγματικά λυπάμαι που βλέπω ότι αυτή η εύθραστη ειρήνη έχει εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή. Μέσω διπλωματικών διόδων θα πρέπει να βοηθήσουμε και απευθύνομαι σε εσά, κύριε Μπορέλ, να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να δείξετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαμεσολαβητή σε αυτή την ενισχυτική κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, Jones. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακόμη μία φορά η πενιχρή αντίληψη της γεωπολιτικής που έχει ο Ντόναλτ Τραμπ ε, έθεσε σε κίνηση μία σειρά από γεγονότα. Δεν φαίνεται να ηρεμούν τα πράγματα, ειδικά μετά την κατάρριψη του Ιρανικού αεροπλάνου. Και συλληπούμε τους ε, συγγενείς των νεκρών. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μπήκε φώτια στην ε, τη αποθήκη και είχαμε έντονες ε, δηλώσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους μεταξύ των οποίων και από τον πρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ΙΠΑ δεν θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Τζόνσον που θέλει να αντικατασταθεί από μια συμφωνία Τραμπ. Ε, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων ανά τον κόσμο, αλλά ειδικά των πιο ευπαθών, που πάντα είναι γυναίκες και τα παιδιά, πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Γκροσέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχουμε ε, αύξηση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια σταθερότητα. Ε, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αόρατη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να επιληθεί η κρίση και να κρατήσει ζωντανή τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Γιατί όποιο και είναι το αποτέλεσμα θα έχει αντίκτυπο σε εμά. Αν υπάρξει κλιμάκωση ε, ή ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα είναι εντός του βεληνικούς των Ιρανικών πυράβλων και θα αντιμετωπίσουμε και μεταναστευτικές ροές αν υπάρξουν ε, περαιτέρω συνομιλίε μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει κατάλληλο ρόλο, γιατί οποιαδήποτε συμφωνία θα έχει συνέπειε στην ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν και η ΕΠΑ θέλουν να είναι σημαντικό προμηθευτή φυσικού αερίου. Αυτό είναι σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για το στόχο μα ε, να είμαστε απελευθερωμένοι από τις εκπομπέ άνθρωποι μέχρι το 2050 και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της στην επίλυση της κρίσης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λίτση, για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, έχουμε μια στάθεια ε, που ξέσπασε λόγω της θανάτου του Και αυτό μας έδειξε την ανεπάρκεια της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, δυστυχώς μιλάμε μόνο για καλή θέληση που δεν είναι αποτελεσματική ούτε έχει συνέπειες στη σημερινή κατάσταση. Κύριε Μπορέλ, αυτά που δεν αφορούν το πρόσωπό σας αφορά το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομικό πλαίσιο. Όμως η ειρηνική οικονομία καταραίει ε, και ε, η κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφου ε, που έχασαν τη 176 άνθρωποι και όλα αυτά μας οδηγούν, καθώς και το περιστατικό με τον Βρετανό πρεσβευτή, όλα αυτά μας οδηγούν σε νέες εντάσεις. Πού είναι η Γεωπολιτική Επιτροπή που μας υποσχέθηκε η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν, με ποιο τρόπο ε, σε αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθήσατε να περιοριστείτε την κλιμάκωση. για το Ιράκ και το Ιράν μιλήσαμε τον Νοέμβριο και ε, συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μειώσουμε τους τόνους και το κάνω και εγώ μέσω της διπλωματίας του διαλόγου και της ανέβρεσης πολιτικής λύσης. Όμως ε, μετά δεν συμβαίνει τίποτα και όλα απλώς καταλήγουν σε μια κοινή δήλωση. Πρώτη δήλωση ε, της κυρίας Φοντερ Λάιεν έφτασε μέρες μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και κόβεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω γιατί έχετε μόλις ένα λεπτό στην διάθεσή σας. Το λόγο τώρα για ένα λεπτό έχει ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν ήταν ε, το θετικό αποτέλεσμα και νίκη μετά από μια υπομονετική διπλωματική προσπάθεια ο πόλεμο τα θύματα και το καθεξής είναι πάντα μια αποτυχία για τη διπλωματία. Γι' αυτό θα πρέπει να, όλο αυτό να εντάσσεται στην ε, γενικότερη στρατηγική μα για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων βάσει τη απλή αρχή ότι είναι πιο εύκολο να αποτρέψουμε κάποιον από το να αποκτήσει τέτοια όπλα παρά να τον πείσουμε να τα καταστρέψει. Όμω, ε, ο Ντόναλντ Τραμπ ε, ακολούθησε διαφορετική οδό σε σχέση με την Βόρεια Κορέα. Επομένω, έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη εδώ στην περιοχή. Ακούμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα τρομοκρατών. Όχι, είναι μια μεγάλη χώρα με 80 εκατομμύρια επικόους, πολύ, με πολύ νεανικό πληθυσμό. Τους ξέρω γιατί ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, των σχέσεων με, την Ιράν, με το Ιράν. Επομένω, ε, υπάρχει ένα ε, τεράστιο φάσμα θετική και ειρηνική συνεργασία που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Μπενιφέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αποκλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ε, μετά από τη μεγάλη ένταση λόγω ε, της δολοφονίας του Σουλεϊμανή είναι Καλή είδηση, όμως ο δρόμος είναι μακρύς. Ε, η Συμφωνία για τα Πυρηνικά οδήγησε στην χώρα στο να είναι εταίρος μας στο διάλογο μετά από πολλά χρόνια θα πρέπει να γίνει σεβαστή η συμφωνία αυτή. Όπως είπατε κύριε είπατε εκπρόσωποι, στο ε, περιθώριο του ε, Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ε, συζητήθηκαν τα θέματα αυτά. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο Ιράν και λόγω των οικονομικών κυρώσεων της Αμερικής. Την τι περασμένε ε, ημέρες επιδεινώθηκε η κατάσταση λόγω και της κατάρριψη ε, του αεροσκάφου ε, Το Ιράν δεν ακολουθεί την οδό της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων που επιθυμούμε και αυτό πρέπει να είναι μέρος του έργου μας και της συνομιλίας μας με τις Ιρανικές Αρχές. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπονφρίσκο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει μια επιθυμία στο στήθος ε, των ε, Ιρανών και των ε, Ιρακινών. Θέλουν να ξεφορτωθούν αυτές τις κυβερνήσεις τους. Θέλουν ασφάλεια, ευημερία και ειρήνη. Και έτσι έχουμε αυτές τις διαμαρτυρίες που βλέπουμε στο Ιράν, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν την αδιαφορία την δική μας και της διεθνούς κοινότητας. Και ήδη έχουν υπάρξει εκατοντάδες νεκροί. Όλα αυτά βεβαίως θυμίζουν το 1979. Και βεβαίως υπάρχουν δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έρχονται από την Ευρώπη για να στηρίξουν ανθρωπιστικά αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν μεγαλύτερο τρομοκράτη ε, όσα συνέβησαν στο Ιράκ και στο Ιράν είναι σχετικά και επικίνδυνα. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασιστικοί. Και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν ξεκάθαρα. Η δολοφονία του στρατηγού Σουλημενή από τη ΣΥΠΑ ε, ήταν μια τρελή πράξη δικαστέα ε, που ενισχύει τους εχθρούς της ε, δημοκρατίας και σήμερα εμεί δεν πρέπει να διαπράξουμε το εξή λάθος, να πετάξουμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά, γιατί είναι ακόμη πιο σημαντική από πριν, όπως είπε και ο υπότος Για μας είναι πραγματική δοκιμασία αυτή. Και τελικά είτε στο Ιράκ ε, είτε στο Ιράν έχουμε μια κοινωνία των πολιτών που ζητά διαφάνεια και ε, δημοκρατική ανάπτυξη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους άνδρες και αυτές τις γυναίκες για να υποστηρίξουμε τη διπλωματική και πολιτική οδό και για να αποφύγουμε κλιμάκωση της έντασης ε, που δεν έχει ακόμη εξελιχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό 1,5 λεπτό. Κύριο Σπίκουλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση του αεροσκάφους ε, στο Ιράν. Στηρίζω τις προσπάθειες των ε, ερευνητών από όλες ε, τις χώρες που έχασαν ε, πολίτες τους ε, σε αυτή την τραγωδία. Το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μονομερείς ενέργειες, γιατί οι συνέπειες ενδέχεται να είναι τόσο σκληρές όσο αυτές που βλέπουμε εδώ. Η δολοφονία του ε, στρατηγού Σολαϊμάνη άνοιξε αυτό το κουτί της Πανδώρας με απρόβλεπτες ε, συνέπειες. Ελπίζω ότι η τελευταία είδηση που ακούσαμε με την απόσυρση των ε, Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ δεν ε, θα αποτελέσει αιτία περαιτέρω συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσει προδραστικά, να ε, προτείνει διπλωματικές λύσεις με στόχο το Ιράν να σεβαστεί όλες τις δεσμεύσεις του που απορρέουν από την Συμφωνία για το Πυρηνικά. Σίγουρα θα πρέπει να σταματήσει η βία από τις Ιρανικές Αρχές προς τους ε, διαδηλωτές που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Και έτσι σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για την διατλαντική συνεργασία στην επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη διαδικασία Catch έχουμε λάβει πολλά αιτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσω τον αριθμό των ομιλητών ανά πολιτική ομάδα. Ξεκινούμε με τον κύριο Σβέρευ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, ακολουθώ τις ε, ε, προσπάθειες της ελληνικής αντιπολίτευσης ε, για δημοκρατία και ελευθερία. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχουμε αφιερώσει την προσοχή μας ακριβώς στην Ιρανική αντιπολίτευση. Ωστόσο, η υπηρεσία εξωτερικής ε, πολιτικής έχει ε, διαφορετική προσέγγιση προς εκείνους. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, με μεγαλύτερο στένος να σταθεί στο πλάι της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και να μην προσπαθεί να διαμεσολαβεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μεταξύ της ε, χώρας ε, της ελευθερίας και μεταξύ της χώρας που έχει σκοτώσει και συνεχίζει να σκοτώνει ε, εκατοντάδες και χιλιάδες πολιτών, διαδηλωτών, καταρρύπτει αεροσκάφη των πολιτικών ευραμών και το καθεξής. Καλό λοιπόν τον κύριο Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναδιαμορφώσει την πολιτική της για το Ιράν. Για ένα λεπτό κύριο E, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά πρέπει να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση και να αποκλιμακώσουμε την ένταση. Είδαμε τον θάνατο του στρατηγού Σουλεϊμανίου ανεξαρτήτως του ποιος ήταν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έτσι κλιμακώθηκε η κατάσταση. Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε επικριτικά προς τις ΗΠΑ. Να είμαστε εταίροι. Αντάξει των άλλων χωρών. Και να καταβάλουμε τέτοιες προσπάθειες έχουμε καλές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και με άλλους, αλλά και με το Ιράν. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την ε, πυρνική συμφωνία, γιατί ε, οποιαδήποτε αύξηση της έντασης και κλιμάκωση στο επίπεδο του πολέμου είναι αντιπαραγωγική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αουστρεβίτσιους έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ιρανικό καθεστώς ε, αξίζει βεβαίως κυρώσεις ε, για τη δράση του κατά του ίδιου του του λαού που βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί αλλά και για τα εγκλήματα πολέμου όπως η κατάρριψη του Ουκρανικού αεροσκάφους. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε κυρώσεις κατά του καθεστώτος και να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση. Όσο παραμένουμε αδρανείς, ε, ενθαρρύνεται το καθεστώς για να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ας παραδεχτούμε τα λάθη που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ιράν, καθώς είχαμε πολύ αισιόδοξε προσδοκίες. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κονέτσινα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει εδώ στο Κοινοβούλιο να συνειδητοποιήσουμε ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι αγώνας ποδοσφαίρου. Δεν θα πρέπει να αγώμαστε όλα τα φάουλ της αγαπημένης μας ομάδας, ε, ενώ καταδικάζουμε την αντίπαλη ομάδα. Το... Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με το διεθνέ δίκαιο. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να ασκούμε κριτική σε οποιονδήποτε παραβιάζει ε, του ε, κανόνε. Ε, στην περίπτωση αυτή, οι Ηνωμένε Πολιτείε αντιμφισβήτητα παραβίασαν το διεθνέ δίκαιο και πρέπει να καταδικάσουμε φυσικά και την κατάρριψη του αεροσκάφου από το Ιράν εδώ δεν είναι το καθήκος μας να υπερασπίσουμε ε, το Ιράν ή να κατηγορούμε τι Ηνωμένες Θα πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς ε, δικαίου. Το 2020 δεν ξεκίνησε καλά και αν δεν αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο διεθνές δίκαιο μπορεί και να μην τελειώσει και καλά. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, αλλά όχι μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν, αλλά μεταξύ του διεθνούς δικαίου και του χάους. Ας διαλέξουμε. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Ουλρίκ, για ένα λεπτό. Καταρχήν, θα ήθελα να παραπονεθώ στο Προεδρείο, γιατί μας έχουν απαγορεύσει να έχουμε σημαίες στην Ολομέλεια. Είναι πραγματικά απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, η συμφωνία για τα πυρηνικά είναι καλό αποτελέσμα της ευρωπαϊκής διπλωματίας, αλλά πρέπει να πούμε ότι κάθε κακό που συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή οφείλεται στην επιθετική πολιτική των ΗΠΑ και κατάφορα αγνοούν το διεθνές δίκαιο. Έχουν διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις κατά πολιτικών άλλων χωρών. Και θέλω να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να καταδικάσει αυτή την τρομοκρατική επίθεση, τον είπα, με τον ίδιο τρόπο που καταδικάζεται τις τρομοκρατικές επιθέσεις άλλων χωρών. Και παρακαλώ να κρατηθείτε μακριά από αυτές τις αιματηρές περιπέτειες στον ΗΠΑ. Ευχαριστώ κύριος Μπασέσκου για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με την Αμερικανο-Ιρανική διένεξη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο στρατηγός Σουλεϊμανή ήταν ένας από τους ε, οργανωτές της επίθεσης ε, κατά της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη και εκτελέστηκε σε Ιρακινό έδαφος εκεί όπου διέπραξε την τρομοκρατική πράξη. Σε ό,τι αφορά εμάς. Υπάρχει ένα γενικό ρεύμα ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά. Θα ήθελα να εκφράσω τη δική μου άποψη. Το Ιράν δεν θα σεβαστεί την Πυρηνική Συμφωνία και εμείς θα μείνουμε αλληλέγγυοι με μια τρομοκρατική εξουσία στην Τεχεράνη. Ας ε, επικεντρωθούμε στην ε, αλληλεγγύη. Δεν ξέρω όμως αν τελικά θα μπορέσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι ως το τέλος ε, όταν μιλάμε εδώ για μια κυβέρνηση τρομοκρατική η οποία είναι τέρους μας σε αυτή την πυρηνική συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για ένα λεπτό. Είπατε εκπρόσωπε Μπορέλ τα 176 θύματα του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από ένα Ιρακινό πύραυλο την περασμένη εβδομάδα είναι τραγική παράπλευρη απώλεια ενό σπιράλ δράσης αντίδρασης. Και όταν γνωρίζουμε ότι οι Ιρακινικές αρχές αναγνωρίζουν την αλήθεια, ε, αφού ε, την ε, δημοσίευσε ο Καναδός Πρωθυπουργό είναι ακόμη χειρότερο. Όμως μπορεί να έχουμε και ακόμα χειρότερα, ε, χειρότερες εξελίξεις. Είχαμε δεκάδες Καναδούς και κάποιους Ευρωπαίους μεταξύ των θυμάτων, όμως Είχαμε και πολλούς Ιρανούς και είχαμε μεγάλη καταστολή με νεκρούς και τραυματίες στο Ιράν, όπως είδαμε και ε, επίσης ε, ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταργηθεί η Συμφωνία για την Πυρηνικά το 2015 αν πρόκειται να ξεσπάσει πόλεμος. Πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε τις διπλωματικές προσπάθειές σας έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχθεί ο πόλεμος αυτός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αλεξάνδρος Φιωρδάνο, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Μπορέλ. Εάν η προσέγγιση της κοινή λογικής δεν επιτυχεί, ε, δεν οδηγεί σε επιτυχία, καθώς και η αποκλιμάκωση, έχουμε άλλα σχέδια δράσης. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Β. Δεν αρκεί να εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας ε, προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, σε ό,τι αφορά τα θύματα λοιπόν του ε, Ουκρανικού αεροσκάφους. Πρέπει να καταστήσουμε σαφέ προ το ελληνικό καθεστώ ότι αν συνεχίσει αυτή την πολιτική στην περιοχή, η απάντηση θα είναι διαφορετική. Και πάλι θα έχουμε μια θύελα της ερήμου. Ο ίδιος ο λαός ε, του Ιράν ε, αντιδρά πολύ πιο έντονα από ότι εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, διαδηλώσεις. Ο αντιμερικανισμός που ακούμε και εδώ, σε αυτή την αίθουσα, δεν ε, απειλεί μόνο τις ΗΠΑ. Αποτελεί απειλή ακόμα και για εμάς εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει και πάλι ο Αντιπρόεδρος και υπότος εκπρόσωπος, ε, κύριος Μπορέλ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ακούσαμε μια σειρά απόψεων, όλες πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ αποκλίνουσες μεταξύ τους. Αν θα έπρεπε να πω σε κάποιον ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας ακούσει αυτή τη συζήτηση, δεν θα ήξερα ποια να διαλέξω. Γιατί πάμε από το ε, απόλυτο λευκό μέχρι το απόλυτο μαύρο. Και αυτό αντανακλά μία κρίση που όπως γνωρίζουμε είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και ενισχυτικό για όλους μας. Ήθελα λοιπόν να πω ότι κανείς δεν εγκατέλειψε την συμφωνία για τα πυρηνικά. Κανείς λοιπόν δεν την έχει εγκαταλείψει. Δεν είμαι εγώ αυτός που θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι ουσιαστική για την ασφάλειά μας και πρέπει να τηρηθεί. Είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών. Και οι τρεις υπουργοί των... της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Γνωρίζω πως ε, υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της επιστολής ε, που μου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που λέει κάτι διαφορετικό από την επιστολή που διάβασα, αλλά για εμένα αυτό το οποίο μετράει είναι η επιστολή που είναι επίσημο έγγραφο και αυτό πρέπει να ακολουθήσω, έτσι. Ο Βρετανός Υπουργός λέει ότι αυτό το οποίο προτείνουν είναι να μην εγκαταλείψουμε την ε, συμφωνία. Και να μην περάσουμε από μια συμφωνία Ομπάμα σε μια συμφωνία Τραμπ. Λέει ότι θέλουμε να διατηρηθεί η συμφωνία ζωντανή. να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός, η διαδικασία, για να έχουμε ένα μοχλό πιέσει απέναντι στο Ιράν. Όχι, όχι. Κανείς δεν έχει εγκαταλείψει την συμφωνία. Η διεθνή Υπηρεσία Ατομική ενέργεια εξακολουθεί να παρακολουθεί, να επιθεωρεί τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν. Και μην ξεχνάμε Η συμφωνία αυτή βεβαίως ε, βασίζεται και σε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χρειάστηκαν 10 χρόνια, δεν είναι κάτι που γράψαμε εμείς μόνοι μας. Και την έχει εγκρίνει και ένα ψήφισμα του ΟΗΕ. Ε, και δεν την έχει ακυρώσει κανείς. Οπότε μην κατηγορείτε εμένα και μου λέτε κύριε Μπορέλ πρέπει να αλλάξετε άποψη. Εδώ δεν σας εξηγώ την άποψή μου. Και αυτήν, εντάξει, αλλά κυρίως τα όσα αποφασίζει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και αυτό το οποίο λέει και η επιστολή των τριών υπουργών. Οπωσδήποτε είμαστε σε επαφή για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν. Και βεβαίως ε, και στο Ιράκ ε, στην διαδικασία των εσωτερικών ε, μεταρρυθμίσεων. Και όταν οι συνάδελφοί μου στο, στο Συμβούλιο Εξωτερικών μου λένε να μιλάω με όλους και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθεί μια περιφερειακή πολιτική λύση. εγώ το βλέπω αυτό ως μια πρόσκληση να είμαι σε επαφή με την κυβέρνηση του Ιράκ. Για την ώρα η κυβέρνηση του Ιράκ είναι υπηρεσιακή, αλλά αμέσως ε, μετά από αυτήν την συνάντηση ήρθα σε επαφή με την κυβέρνηση του Ιράκ ε, και ας είναι υπηρεσιακή. Και την Δευτέρα είχε έρθει εδώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράκ για διαβουλεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και συμφωνήσαμε να κάνουμε περισσότερα και κάποιος με ρώτησε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ναι, το να αναπτύξουμε την ε, συμφωνία σύνδεσης ε, που υπογράψαμε και κυρώθηκε και ενισχύει το 2018. Ναι, το να κάνουμε αυτό, αυτό και μόνο, είναι κάτι σοβαρό ανοίγει σοβαρέ δυνατότητε. Έχουμε μια αποστολή εκεί την οποία μπορούμε να ενισχύσουμε. Η συμφωνία σύνδεση ανοίγει την πόρτα σε σχέσει οικονομικέ, εμπορικέ, ασφαλεία και οπωσδήποτε πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από την σκοπιά της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής με την αποστολή που έχουμε εκεί. Και το λογικότερο θα ήταν να την ενισχύσουμε. για να μην διαλυθεί η χώρα. Γιατί ε, αφού μιλήσατε αντιλαμβάνουμε ότι όλοι γνωρίζετε τις δραματικές συνέπειες ε, που θα έχει για την ασφαλειά μας το ενδεχόμενο μιας κρίσης ε, ανάλογης με αυτήν που βλέπουμε στην Συρία. Γι' αυτό τις επόμενες εβδομάδες και μέρες ε, θα είμαι σε επαφή με τους Ιρακινούς να προσφέρω την στήριξή μας και τη βοήθειά μας για να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη χώρα αυτή και για να μην χαθεί όλη η πρόοδος ε, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά για το ποιο θα είναι το μέλλον, αλλά για την ώρα ένα είναι σαφές το Ιράν δεν είναι σήμερα μια πυρηνική δύναμη χάρη στην συμφωνία αυτή. Και δεν βλέπω πώς μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική συμφωνία. Πραγματικά δεν το βλέπω. Όλοι μιλάνε για αυτή τη συμφωνία. Κάποιοι από εσά ρίξατε και